στην εκλογή του Προέδρου. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού, οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την συμφωνία των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν υπογραφεί είτε από μια κοινοβουλευτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 40 βουλευτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό έχω λάβει τι εξή υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κυρίου Γερζι και της κυρίας Εύα Μπριτ Σβένσον. Οι υποψήφοι μου ανακοίνωσαν πως συμφωνούν με τις υποψηφιότητες του. Οι δύο υποψήφοι θα κάνουν τώρα από μια σύντομη παρουσίαση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την κυρία Εύα Μπριτ Σβένσον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι με στήριξαν κατά τη διάρκεια αυτής της ε, διαδικασίας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη η οποία ε, με έκανε να νιώσω ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ και όλοι μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών που μας απέστειλαν εδώ και να οικοδομήσουμε μια πραγματική Ευρώπη των πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοκρατία ε, εξέφρασε θα έλεγα μέσω αυτού του αποτελέσματος του εκλογικού τις επιθυμίες των πολιτών μας. Αλλά για να είναι λειτουργική, για να είναι πραγματική η δημοκρατία χρειάζεται κάτι περισσότερο από μία απλή έστω και καθολική ψηφοφορία. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση. Συνεπώς θα πρέπει όλοι τώρα να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται γύρω από τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων επιδεικνύοντας φυσικά και τη διαφάνεια η οποία απαιτείται σε διαδικασίες τις οποίες συνήθως ακολουθούμε όπως τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης σαν παράδειγμα. Βιώνουμε όλοι και κυρίως οι συμπολίτε μας μια μεγάλη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση με σημαντικές συνέπειες στον τομέα της απασχόλησης. Ταυτόχρονα βιώνουμε και μια κρίση συνέπεια των κλιματικών αλλαγών η οποία και αυτή η κρίση χτυπάει πριν από ουσδήποτε άλλους τους φτωχότερους του πλανήτη. Η αδικία λοιπόν και η έμβια εξακολουθούν να υπάρχουν σε μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να είμαστε μυρολάτρες. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολιτικές απαντήσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν σε αυτά τα προβλήματα. Οι πολιτικές τις οποίες δυστυχώς ακολουθήσαμε μέχρι τώρα δεν έχουν βοηθήσει να βρεθεί μια λύση. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν όξυναν τις κρίσεις τις οποίες βιώνουμε. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια διαφορετική πολιτική απάντηση. Θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στον Ευρωπαίο πολίτη έτσι ώστε να γίνει η Ευρώπη πιο κοινωνική θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα πρέπει να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, η έμβια. Και κυρίως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική στην οποία να μπορούν να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, να νιώθουν ότι μπορούν να συμμετέχουν. Μια πολιτική δράση η οποία να μην αποκλείει κανέναν να μην αποκλείει κανέναν και ιδιαίτερα ε, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λόγω αναπηριών, λόγω του ε, γενετησίου προσανατολισμού τους κτλ. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στην πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολιτική η οποία θα πρέπει να έχει σαν βασικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα των λεγόμενων των πράσινων, δηλαδή με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι θέσεις αυτές εργασίας όχι μόνο είναι απαραίτητες, αλλά θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν να συνεισφέρουν στην αποτροπή περαιτέρω κλιματικών αλλαγών οι οποίες θα είναι πάρα πολύ αρνητικές για τον κόσμο μας. Επιθυμούμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες της πλήρως. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα πρέπει να προσπαθήσει να δράσει στην διεθνή σκηνή μέσω της σωστής πολιτικής της. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να ακολουθήσει πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης και της χορήγησης ασύλου δίκαιες. Μια ευρωπαϊκή πολιτική χωρίς διακρίσεις, μια Ευρώπη πολυεθνική μια Ευρώπη στην οποία μπορούν να καθρεφτίζονται και να ταυτίζονται μαζί της όλοι οι κάτοικοι της σήμερα και όλοι οι πολίτες. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να σέβεται πριν από οτιδήποτε άλλο τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί πολύ συχνά παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από το που συμβαίνει στον κόσμο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να αποδεχθούμε να κάνουμε συμβιβασμού σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία ήταν και πρέπει να συνεχίσουν να είναι τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαραβίαστα. Και αναφέρομαι εδώ και στην ελευθερία έκφρασης και στα πολιτικά δικαιώματα κτλ. Όλα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν πρέπει να μείνουν απαραβίαστα και βασική ευθύνη συνάδελφοι για όλους μας είναι να τα υπερασπιστούμε οπουδήποτε παραβιάζονται στον κόσμο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πρόσφατα πήραμε την πληροφορία από τον πρόεδρό μας ότι στις εκλογές του μηνός Ιουνίου, τις ευρωεκλογές του μηνός Ιουνίου, το ποσοστό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκε αρκετά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου ε, με ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί αυτό θα βοηθήσει να γίνουν καλύτερα σεβαστά τα δικαιώματα των γυναικών. Ας κάνουμε λοιπόν και άλλο ένα βήμα, ένα βήμα περαιτέρω. Ας προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την επιρροή των γυναικών και στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά και για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα προς το Κοινοβούλιο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν από κοινού να αποδείξουμε στους συμπολίτε μας ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν με αποφασιστικότητα και να σεβαστούμε τις βασικές αρχές μιας πολυπολιτισμικής και πλουραλιστικής κοινωνίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι σας και ο καθένας από εσά μπορεί να επηρεάσει κάπως τα πράγματα. Όλοι έχουμε την δυνατότητα σήμερα να αποστείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα στους συμπολίτες μας, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε την Ευρώπη των πολιτών, θέλουμε την κοινωνική Ευρώπη των πολιτών, θέλουμε να αποδείξουμε στους συμπολίτε μας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα προπαρασκευασμένη να αναλάβει τις ευθύνες της στον τομέα της παγκόσμιας δικαιοσύνης, στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως να αναλάβει τις ευθύνες της σφαιρικές, θα έλεγα πλανητικές ευθύνες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή είναι μια δυνατότητα που έχουμε σήμερα και από εδώ και πέρα για κάποια χρόνια να επηρεάσουμε τα πράγματα. Και αυτό περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστούμε κυρία Σβένσον, αγαπητοί συνάδελφοι. Μου λένε πως ο θόρυβος ε, τον οποίο ακούτε προέρχεται από τον κλιματισμό ο οποίο λειτουργεί γιατί έχουμε τόσο κόσμο και στην αίθουσα και στα θεωρία. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Γκέρζι Μπούζεκ να λάβει τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπούζεκ. Κυρίε και κύριοι, Επίτροποι, εκπρόσωποι του Συμβουλίου θα πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ. Εκπροσωπούμε μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίων και τώρα να σας πω δύο λόγια τον εαυτό μου. Προέρχομαι από τον κλάδο των θετικών επιστημών και το 1980 άρχισα τις ε, επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Αυτό ήταν στο Συνδικάτο Αλληλεγγύη. Εκεί άρχισα να δουλεύω. Μιλούμε για αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη για τον κόσμο, αλληλεγγύη για τα πολιτικά δικαιώματα, αλληλεγγύη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί δώσαμε τη μάχη επομένω για όλα αυτά τα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο πάντοτε ε, αποτελούσε την προσήλωσή μου, αποτελούσε το πιστεύω μου. 97 έως 2001 ήμουν πρωθυπουργός. Και επί μία θητεία τεσσάρων ετών, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να διαπραγματευτούμε την ισότητα τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν εργάστηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην υπηρεσία για νέε τεχνολογίε, καινοτομία και ενεργειακή ασφάλεια. Επίση, ε, ασχολήθηκα και με την αλλαγή του κλίματος, κατά το οποίο απασχόλησε, με ενδιαφέρει. Επίσης ασχολήθηκα και με την πολιτική εταιρικών σχέσεων ε, με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπη. Σε όλους αυτούς τους τομείς εγώ θεώρησα ότι ε, πρόκειται για θέματα προτεραιότητα για την επόμενη εντολή και βέβαια τελικά φτάσαμε τώρα σε μια συγκυρία χρηματοπιστωτική κρίση, μια κρίση που κάνει του Ευρωπαίου να ενατενίζουν προ εμά για να βρούμε μια λύση. Γι' αυτό και θα πρέπει και εμεί να βελτιώσουμε την απόδοση και επίδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο ε, το έχουμε ήδη καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Όμω θα πρέπει να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα ε, και αυτό θα γίνει μόνο εάν τελικά βαδίσουμε με την συνθήκη της Λισαβόνας η οποία θα έχει περάσει από την διαδικασία της επικύρωσης. Ε, μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε στην διεθνή σκηνή. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην ε, πολιτική μας προς Ανατολάς, προς ε, τη Μεσόγειο, προς τις ΕΠΑ, προς τις αναδυόμενες νέες δυνάμεις. Αυτές είναι οι προκλήσεις που μας περιμένουν και γι' αυτό και η συνθήκη της Λισαβόνας νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ εξαιρετικό, πάρα πολύ αξιόλογο με το οποίο μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Τώρα, θα πρέπει να σα αναφέρω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του, του, του έργου μας είναι το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Γιατί πρόκειται για μια κρίση ε, έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτό, να το αναγνωρίσουμε, διότι θα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση. Ε, πολλές φορές οι πολίτες δεν μας καταλαβαίνουν, άρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να μπορούν να μας καταλάβουν καλύτερα, διότι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο θα δουλεύουμε συνέχεια. Ε, όμως το τέλος της εβδομάδας πηγαίνουμε πίσω στην πατρίδα μας και εκεί θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση του έργου μας εκ μέρους των πολιτών να καταλάβουν ότι κάνουμε αυτό το οποίο περιμένουν από εμά. Και έτσι θα είναι πιο εύκολο να επιτελέσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Γκέρζι Μπούζικ. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού, σας υπενθυμίζω πως για να εκλεγεί ένας ή μία υποψήφιος θα πρέπει στους τρεις πρώτους γύρους των ψηφοφοριών να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των καταμετρημένων ψήφων. Σοβέλτια που δεν έχουν συμπληρωθεί ή είναι άκυρα δεν θεωρούνται καταμετρημένες ψήφοι. Τώρα τυχαία θα επιλέξουμε 8 καταμετρητές ψήφων. Theo Karous. Der Kollege da, der Kollege Theo. Είναι εδώ ο συνάδελφος. Ja, Herr... Ωραία. Κυρία συνάδελφε, με συγχωρείτε, έχω εδώ πέρα μόνο το όνομα δεν γράφει αν είστε κυρία ή κύριος. Είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε αυτή την ευθύνη. Ωραία. Ευχαριστώ. Andres Barea. Andres Barea. Frau Kollegin, sind Sie... Κυρία συνάδελφε, Είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε αυτή την ευθύνη. Ευχαριστώ. Ούτε η πρώην Υπουργοί Εξωτερικών γλιτώνουν. Κύριε Σέβεριν, είστε διατεθειμένος να αναλάβετε αυτή την ευθύνη, θαυμάσια. Jetzt, Frau Kollegin oder Herr Kollege Hübner. Hübner. Hübner. Frau, ah, dann Η συνάλφος Χίμπνερ. Α, με συγχωρείτε. Το έχουν γράψει αλλιώ το όνομά σας από ότι είναι κανονικά. Ωραία, λοιπόν, η κυρία Χίμπνερ. Οπότε τώρα ο συνάλφος Κορ, Δίτερ Κοχ... Δεν βλέπω να υπάρχει άλλο συνάλφος με αυτό το επώνυμο, οπότε είναι ο Ντίτερ Κοχ. Και τώρα η συνάλφος Head λοιπόν. Head. Ανά Head. Θα αποδεχτείτε αυτή την ευθύνη. Βλέπω μεγάλη χαρά. Ναι. Ja, Ναι, και οι πρόεδροι των ομάδων, κυρία Ρεμπέκα Χαμ, είστε διατεθειμένοι να το κάνετε αυτό ωραιότατα, με χαμόγελο. Και τώρα, Ματ λένε ο συνάδελφος ή η συνάδελφος Ματλένε, ποιος είναι Α, ο κύριος Ματλένε και εσείς δέχεστε οπότε έχουμε 8 καταμετρητές ψήφων πρέπει να ξαναπώ τα ονόματα ναι, σύμφωνα με τον κανονισμό ωραία Θα λέω τα ε, επώνυμα, πέρα γιατί δεν έχω πλήρω τα ονόματά σας. Η κυρία Λαρούς είναι για τα ονόματα Α έως Β, Μπαρέα για την κάλπη C έω E στο λατινικό αλφαβητό. Σεβερίν για τα γράμματα F έω H κυρία Χίμπνερ για τα γράμματα I έως K, συνάδελφο Κόχ για τα γράμματα L έως M, η συνάδελφος Χέιτ για τα γράμματα N έως R, Harms για το γράμμα S και Ματλένο για το γράμμα TAF έως Z. έχετε, σας έχουν μοιραστεί οδηγίες για την εκλογή του Προέδρου. Θα μοιράσουμε τώρα τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους. Τώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού μας, θα περάσουμε στην εκλογή του Προέδρου. Έχετε ήδη ψηφοδέλτια και φακέλους. Ωραία, παρακαλώ λοιπόν να βάλετε ένα σταυρό στο τετραγωνάκι δίπλα στο όνομα του ή της υποψηφίου που επιλέγετε. Μπορείτε να ψηφίσετε έναν μόνο. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτό το οποίο ψηφίσετε, ζητήστε από έναν κλητήρα ένα νέο ψηφοδέλτιο. Ο κλητήρας θα σας δώσει ένα νέο ψηφοδέλτιο και θα πάρει από εσάς το λάθος συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο το οποίο θα καταστραφεί. Οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό σημάδι ή καταχώρηση ή ψήφος σε πάνω από ένα άτομα καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο. Παρακαλώ διπλώστε το δύο φορές και βάλτε το στον φάκελο και ψηφίστε στην κάλπη που αντιστοιχεί στο όνομά σας σύμφωνα με το λατινικό αλφάβητο όπως τα διάβασα. Δεν θα σας καλέσουμε να ψηφίσετε ονομαστικά. Εγώ θα περιοριστώ στο να κηρύξω την έναρξη και το πέρας της ψηφοφορίας. Επειδή τα ονόματα των βουλευτών που ψηφίζουν με μυστική ονομαστική ψηφοφορία πρέπει να εμφανιστούν, θέλω να σας παρακαλέσω να υπογράψετε στον κατάλογο που υπάρχει πριν πάτε στις κάλπες. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω πως θα πρέπει να ρίξετε στην αντίστοιχη κάλπη τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο και θα ήθελα να σας πω εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να δείξετε στους καταμετρητές των ψήφων την ταυτότητά, την ταυτότητά σας. Οι ίδιοι καταμετρητές των ψήφων θα ψηφίσουν στο τέλος. Σας παρακαλώ λοιπόν να κατευθυνθείτε στις κάλπες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 Could to the for A to B, please? Κυρία Τέο Κάρος, η οποία καταμετρά τους ψήφους θα μπορούσε να έρθει στην κάλπη για τα γράμματα Α και Β. Ευχαριστώ.